που είναι πολύ σημαντική ε, για την προσέλκυση των ξένων επενδύσεων. Όλα δηλαδή είναι στα χέρια μας, είναι στο χέρι μας να έχουμε αποτελέσματα. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώνω τη συζήτηση για το θέμα αυτό. Η ψηφοφορία θα λάβει χώρα αύριο στις 12.30. Προχωρούμε στην έκθεση του κυρίου Μίλοσλαβ Ράνσντορφ «Εμπορικές πτυχές της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης». Θα ήθελα να ξεκινήσω δίνοντας το λόγο στον εισηγητή για τέσσερα λεπτά. Παρακαλώ. Έχετε το λόγο για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στους αγαπητούς συναδέλφους και στους εκπροσώπους της Επιτροπής για την συμμετοχή τους στη συνεδρίαση αυτή. Θα σας πω τι ακριβώς ε, εννοώ στην ε, έκθεση αυτή. Στόχος είναι η πρόθεση και η ενδυνάμωση του κράτους δικαίου και της κοινωνίας των πολιτών στις χώρες ε, της Ανατολικής Σύμπραξης. Συνεργαζόμαστε από κοινού, συνεργαστήκαμε και προετοιμάσαμε 142 τροπολογίες και με αυτόν τον τρόπο μπορέσαμε να υποβάλουμε και μερικές ε, τροπολογίες ε, συμβιβασμού. Την τελευταία στιγμή οι συνάδελφοι της Ολμάδας Σοσιαλιστών και Δημοκρατών συνέταξαν δύο προφορικές τροπολογίες. Ο κύριος Κούτες, εξ ονόματος των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, υπέβαλε δύο τροπολογίες, όπως σας είπα, που τις αποδέχομαι, δεν έχω κανένα πρόβλημα να δεχτώ τις δύο αυτές τροπολογίες και θα σας εξηγήσω για ποιο λόγο γιατί η σε βάθος και σφαιρική ζώνη ελευθέρων συναλλαγών είναι πάρα πολύ σημαντική σε αυτή την οικονομική περιοχή και περιοχή συναλλαγών. Θα μπορούσα όμως να αναφέρω και άλλες στρατηγικές για άλλε εμπορικέ στρατηγικέ. Είμαι συνεπώ υπέρ αυτή τη πρόταση, παρόλο που βεβλήθη την τελευταία στιγμή. Σε ό,τι αφορά τη γεωργία. Η γεωργία είναι ένα άλλο θέμα. Η πρόταση του κυρίου κουτά εξ ονόματος Σοσιαλιστών και Δημοκρατών η Γεωργία έχει ε, κατηγορηθεί για παραβίαση δικαιωμάτων των παιδιών, χρησιμοποιείται δηλαδή εργασία ανηλίκων, ενδεχομένως ε, δεν έχουμε στοιχεία για την καταγγελία αυτή, αλλά η προστασία των δικαιωμάτων των ανηλίκων είναι η παριθμόν ένα προτεραιότητά μου. Δεν έχω λοιπόν κανένα πρόβλημα να δεχτώ αυτή την προφορική τροπολογία που υπέβαλε ο κύριος Κούτας. Θα ήθελα όμως να αναφέρω ότι ο πρόεδρος της Γεωργίας, ο κύριος Σούλη, είναι ένας πολύ καλός φίλος των ΗΠΑ ένας ε, σεβαστός δημοκράτης, ο οποίος έγινε δεκτός εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ενδεχομένω θα θυμάστε όταν ε, έλαβε το λόγο εδώ στο αυτό το Κοινοβούλιο. Αυτά λοιπόν ως προς την έκθεση αυτή. Θα ήθελα να πω επίσης ότι οι κοινοβουλευτικέ παρεμβάσει θα πρέπει να είναι σαν τις φούσε των γυναικών, αρκετά μακριέ για να καλύπτουν το θέμα και αρκετά ε, κοντές για να μην προκαλούν. Ξέρω ότι δεν κατάφερα να επιτύχω αυτό τον ιδανικό στόχο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Ράνστορφα. Περνάμε τώρα στο Catch the Eye. Ε, μας έχουν υποβληθεί τέσσερα αιτήματα. Να ξεκινήσουμε από τον κύριο Μιγκάλσκι. Ε, Κυρίες και κύριοι, είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που μας δίνει τη δυνατότητα να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Υπάρχουν πάρα πολλά αξιόλογα στοιχεία σε αυτή την έκθεση. Υπογραμμίζουμε το γεγονός ότι η Ευρώπη εξέφρασε την αντίρρησή της σε αυτές ε, τις διαπραγματεύσεις. Αυτό θα έχει πάρα πολύ αρνητικές επιπτώσεις. Υπάρχουν και ορισμένες πληροφορίες που αφορούν τις διάφορες χώρες. Ορισμένες χώρες όπως η Γεωργία για παράδειγμα, όπως τη Γεωργία για παράδειγμα, η κατάσταση είναι καλύτερη. Σε άλλες χώρες όπως η Ρωσία η κατάσταση είναι λιγότερα καλή. Αυτό μας προβληματίζει ιδιαίτερα. Είναι σημαντική παρόλα αυτά αυτή η συνεργασία παράλληλα με την πολιτική και κοινωνική συνεργασία. Αυτό θα πρέπει να το υπογραμμίσουμε. Αυτό μετράει ιδιαίτερα το να υπάρξει συνεργασία με αυτές τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Ευχαριστώ πολύ. Κύριο Τικάου. Η κυρία Τικάου. Ε, ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα που συζητάμε. Με χαροποιεί η πρόσβαση της Μολδαβίας σε αυτή τη συμφωνία γιατί αυτό θα βοηθήσει την Ένωση να επιτύχει τους στόχους για την ενέργεια και την ασφάλεια και θα συμβάλλει στην ενέργεια και στην ασφάλεια αυτών χωρών. Θα επιθυμούσα να υπάρξει συνεργασία σε αυτό το τομέα με την Ουκρανία και αυτό θα δώσει τη δυνατότητα να ξεκινήσουν κοινά προγράμματα για, για ε, ε, που θα αφορούν τι υποδομέ. Θα ήθελα να ζητήσω από την Επιτροπή να ξεκινήσει μια στρατηγική για την περιοχή τη Μαύρη Θάλασσα, γιατί παίζει σημαντικό ρόλο στην πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Μαύρη Θάλασσα έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο δυναμικό για τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργεια. Ο κύριος Σεκέρσκι παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, είναι σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει τη στήριξη της στις χώρες αυτές. Θα πρέπει να συμβάλλουμε έτσι ώστε να επιτευχθεί μια πολιτική και οικονομική ενοποίηση για αυτές τις χώρες στα πλαίσια της συνεργασίας μαζί τους και κυρίως με βάση τα πλεονεκτήματα που θα έχει η οικονομική συνεργασία. Η Ευρώπη διανύει μια περίοδο κρίσης και θα πρέπει να δημιουργήσει μια νέα στρατηγική για τις χώρες μέλη του Νότου. Σε αυτό το πλαίσιο

Ε, είναι καλό να υπάρξει η απελευθέρωση του εμπορίου με αυτές τις χώρες και αυτό πρέπει να είναι φυσική απόρρια της πολιτικής συνεργασίας. Αυτό θα παίξει μεγάλο ρόλο για την οικονομική ανάκαμψη, τις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις αλλά και την ασφάλεια της ενέργειας. Πάνω σε αυτή τη βάση καλό την Κομισιόν να παρουσιάσει κατεπηγόντως την στρατηγική για τον εύξηνο πόντο και υπογραμμίζω τη σημασία των ε, χωρών ε, διαμετακόμισης. Η Ρουμανία είναι πολύ ε, δραστήρια εδώ. Κάναμε ένα πρόγραμμα για τη μεταφορά μέσω της γεωργίας του αερίου ε, και από τον Εύξηνο Πόντο. Επίσης έχουμε συνεργασία και με τη Μολδαβία, ε, αγωγούς αερίου, ε, μεταφοράς ηλεκτρικού για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση εκεί. Ο τελευταίος ομιλητής είναι ο κύριος Πασκά. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, κύριε Πρόεδρε, όταν μιλάμε για την ανατολική εταιρική σχέση, συχνά προσπαθούμε να δώσουμε μαθήματα στους εταίρους μας, πώς, θα, πώς να διαχειριστούν τις χώρες τους. Όμως ε, η οικονομική δυναμική της συνεργασίας ε, πολλές φορές δεν ενεργοποιείται. Η Ουκρανία είναι ο πιο σημαντικός ανατολικός γείτον και, είναι, και το, το άνοιγμα της συνεργασίας ε, θα μπορούσε να βελτιώσει τα οικονομικά μας δεδομένα. Καλό θα ήταν λοιπόν να ξεπεράσουμε τα προβλήματα με τις θεωρήσεις γιατί έτσι πολλοί Ουκρανοί θα ήταν διατεθειμένοι να έρθουν στο νότο της Ευρώπης, να πάνε στην Ιταλία ή την Ισπανία και σίγουρα θα ήθελαν και ως τουρίστες να επισκεφθούν τις χώρες αυτές, πράγμα το οποίο θα δημιουργούσε θέσεις εργασίας σε αυτές τις περιφέρειες της Ευρώπης. Από την άλλη πλευρά, επειδή ε, είναι ε, καλή η θέση των μεσαίων στρωμάτων, είναι ισχυρή η μεσαία τάξη στην Ουκρανία, θα μπορούσαν να αγοράσουν ευρωπαϊκά προϊόντα. Αλλά υπάρχουν πολλά εμπόδια και δεν έχουν πρόσβαση στα προϊόντα αυτά. Αυτά τα εμπόδια πρέπει να καταρρύψουμε για να στηρίξουμε το εμπόριο. Το εμπόριο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και για να κλείσουμε τη συζήτηση να δώσω το λόγο στον Επίτροπο Καλάς. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, είναι χαρά μου που μπορώ να συζητήσω μαζί σας την εμπορική πολιτική της Ευρώπης προς τους ανατολικούς γείτονες. Ευχαριστώ τον κύριο Ράνστορφ, τον εισηγητή που ανέλαβε την πρωτοβουλία για την έκθεση αυτή αλλά και όλα τα αξιότιμα μέλη που συμμετείχαν στην επικοδομητική συζήτηση επί του κειμένου καλύπτεται όχι μόνο το εμπόριο στα αγαθά αλλά και συνεργασία σε άλλους συναφείς τομείς όπως προστασία του, των επενδύσεων, ε, εξυγχρονισμός, ε, κατάρρευση ε, μη τελωνιακών εμποδίων κλπ. Όπως ξέρετε, τον τελευταίο μήνα υπήρξαν ιδιαίτερα σημαντικές εξελίξεις για τις εμπορικές σχέσεις με τους περισσότερους ανατολικούς γείτονες οι διαπραγματεύσεις για αυτήν την ζώνη ελευθέρων συναλλαγών DCFTA, βαθιά και συνεκτική, ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο και τα δύο μέρη προτίθεται να συνεχίσουν και να προχωρήσουν στην μονογράφηση του κειμένου της DCFTA στις 16 Ιουλίου όταν γίνει η εξέταση του κειμένου και οριστικοποιηθεί. Τώρα η Ουκρανία θα πρέπει να δημιουργήσει συνολικές πολιτικές συνθήκες που θα, θα επιτρέψουν την ε, υπογραφή και την ε, ε, επικύρωση. Είναι πολύ σημαντικό ε, λοιπόν να ε, εγκριθούν η, να εγκριθεί η DCFTA πριν από τη Συμφωνία Σύνδεσης και πριν ε, αποφανθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το πρώτο εξάμεινο φέτος βελτιώθηκαν οι διμερείς σχέσεις με Μολδαβία, Γεωργία, Αρμενία, τρεις εταίρους όπου οι διαπραγματεύσεις ε, στα πλαίσια του DCFTA άρχισαν προχώρησαν και καλά οι διαπραγματεύσεις χάρη στην διεξοδική προπαρασκευαστική διαδικασία των περασμένων ετών. Είναι σημαντικό ότι άρχισαν οι μεταρρυθμίσεις και τώρα πρέπει να συνεχιστούν. Οι διαπραγματεύσεις στα πλαίσια του DCFTA είναι η αρχή μιας μακράς διαδικασίας μεταρρυθμίσεων. Με την Λευκορωσία και το Ατζερμπαϊτζάν η Κομισιόν θα ακολουθήσει παρόμοια ατζέντα όπως και με τους άλλους ανατολικοευρωπαίους εταίρους. Η Κομισιόν όμως πιστεύει ότι η συμμετοχή στον ΠΟΕ και οι βασικές μεταρρυθμίσεις στο εμπόριο και στις άλλες εμπορικές ε, ε, πτυχές της οικονομίας αυτών των χωρών εταίρων είναι σημαντικό για να βελτιωθεί και η εμπορική μας ατζέντα. Για να αρχίσουν διαπραγματεύσεις ε, με την Κομισιόν θα πρέπει οι εμπορικοί εταίροι να έχουν την ικανότητα να εφαρμόσουν την DCFTA. Δυστυχώς το Αζερβαϊτζάν και η Λευκορωσία τώρα δεν συμμορφούνται προς τις ε, προϋποθέσεις αυτές και δεν διαθέτουν την αντίστοιχη ικανότητα. Θα πρέπει να τονίσω ότι οι διμερείς εμπορικέ σχέσεις μας με τους ανατολικοευρωπαίους εταίρους δεν μπορεί να αποσυνδεθούν από το ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούν. Αυτό το μήνυμα ισχύει παντού για όλους τους εταίρους μας. Θέλω να καταγράψω ότι αυτό ευθυγραμμίζεται και με τις βασικές αρχές της ανατολικής εταιρικής σχέσης ε, σύμφωνα με την οποία το DCFTA, τα DCFTA αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των ε, συμφωνιών σύνδεσης και δεν μπορούν να ειδωθούν απομονωμένα. Ε, ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, η Λευκορωσία συμμετέχει στην πολυμερή διάσταση της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, θεωρώ ότι συνολικά η έκθεση που ετοίμασε ο εισηγητής κ. Ράνστορφ αντικατοπτρίζει σωστά το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Κομισιόν συμμερίζονται τις ίδιες απόψεις επί των εμπορικών σχέσεων με τους ανατολικούς μας εταίρους. Ε, είναι πολλές οι τροπολογίες που προτάθηκαν και από την άλλη βλέπω ότι υπάρχει μεγάλη υποστήριξη της έκθεσης. Αυτό δείχνει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει δεσμευτεί να προωθήσει περισσότερο τις διμερείς εμπορικές σχέσεις με τους ανατολικούς, ε, ανατολικοευρωπαίους εταίρους. Χαιρετίζω και την ε, κοινοβουλευτική συνέλευση Euronest που είναι πολύ σημαντική. Σας διαβεβαιώνω ότι η Κομισιόν συμφωνεί απόλυτα επί της ανάγκης να προωθηθεί μια φιλόδοξη εμπορική ατζέντα ως καταλήτης μεταρρυθμίσεων για τους ανατολικοευρωπαίους εταίρους και δείχνει την προθυμία μας να προωθήσουμε αυτή την ατζέντα. Ε, βέβαια, το καθήκον δεν θα είναι εύκολο. Θα πρέπει να είναι σημαντικό να συνεχίσει η Κομισιόν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συνεργάζονται στενά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ολοκληρώνεται η συζήτηση. Ψηφοφορία θα λάβει χώρα αύριο στις 12.30. Περνάμε τώρα στο τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Θα συζητήσουμε την